Συνάδελφοι, σας παρακαλώ καθίστε. Παρακαλώ, κοιτάξτε, φροντίστε να έχετε όλοι τις κάρτες, τις ηλεκτρονικές για την ψηφοφορία. It's too Λοιπόν, συνάδελφοι, μαραθώνια ψηφοφορία σήμερα. Με ακούτε όλοι καλά. Λοιπόν, ψηφίσουμε. Πρώτη έκθεση, ένσταση Σήμερα το πρωί είχαμε την ανταλλαγή απόψεων, ο συνάδελφος Καρλ Σλούτερ και η κυρία Ρενάτε Ζόμερ ζήτησαν μαζί να γίνει μια τροποποίηση στον κατάλογο ψηφοφορίας και να ψηφίσουμε σε μπλοκ. Υπάρχουν αντιρρήσεις για αυτό, για αυτή τη διαδικασία, να ψηφίσουμε δηλαδή κατά μπλοκ. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Άρα έτσι και θα ψηφίσουμε. Πρώτο μπλοκ. Πρώτη ομάδα. Προτείνω να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Κρίς, ναι, μπορείτε να διευκρινίσετε... Είπατε η πρώτη ψηφοφορία ε, on block δηλαδή. Το πρώτο μπλοκ Επαναλαμβάνω. Το πρώτο μπλοκ περιλαμβάνει τις αιτιολογικές σκέψεις 4 έως 8. Έπειτα, το επόμενο μπλοκ, αιτιολογικές σκέψεις B μέχρι H, μέχρι I, με συγχωρείτε, και στο τρίτο μπλοκ ψηφίζουμε για την παράγραφο 3 και 4. Και τέλος η συνολική ψηφοφορία. Άλλες ερωτήσεις? Ήταν τελευταία στιγμή αυτή η πρόταση, γι' αυτό σας ρωτώ αν υπάρχουν αγιοτήρεις. Ψηφίζουμε το πρώτο μπλοκ, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Περιμένω. Ψηφίσατε όλοι. Haben alle abgestimmt. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται το πρώτο. Μπλοκ, πάμε στο δεύτερο. Αιτιολογικές σκέψεις B μέχρι I. Η ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται και αυτό. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε για τις παραγράφους 3 και 4 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται επίσης. Τώρα, τελική ψηφοφορία, όπως έχει τροποποιηθεί, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. «28 ψήφοι υπέρ 27 κατά μία αποχή εγκρίνεται για μία ψήφο». θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο και εκεί χρειάζεται ενισχυμένη πλειοψηφία. Περνάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Ένσταση πολλών συναδέλφων για του έλεγχου στα προϊόντα ζωική πρόέλευση. σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφο 2, ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 42 υπέρ, 18 κατά, 2 αποχές, εγκρίνεται. Αυτά ήταν τα εύκολα. Πάμε στα δύσκολα τώρα, στη μαραθώνια ψηφοφορία, έκθεση Ροτ Μπέρεντ. Αρχίζουμε λοιπόν. Unblock. 222-223 υπέρ. 224. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.24-2.25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 2.28. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. ε, περισσεύει ένα μέλος των σοσιαλδημοκρατών. Ένα συνάδελφος περισσεύει τώρα. Είμαστε εντάξει πέρας. 38 προς 26 εγκρίνεται. 2,29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2,30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση 230. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 240. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 2.39 ε, αποσύρθηκε. 2.42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 243. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές η ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.44 και 2.43 είναι ταυτόσιμες. Ήμκο 18 καταπίπτει, 246 και Ήμκο 19 υπέρ. Κατά. Αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση, 246 και Ήμκο 19, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνατε. Ενοποιημένη τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.52. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 252. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 35 υπέρ, 28 κατά, εγκρίνεται. 2,55 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 253 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 256 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 257 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 258 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές ηλεκτρονική επαλήθευση. 258. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 259 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 261 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 261. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Ήμκο 23. Υπέρ. Κατά. Μόνο 15 ψηφίζεται. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ήμκο 23. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται, σαφέστατα. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υποθέτω πως εγκρίνεται. Θα κοιτάξουμε επαλήθευση ηλεκτρονική. 25. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ήμκο η 24 καταπίτη 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 29. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.64 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 263 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται, λέτε, ηλεκτρονική επαλήθευση. 263. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 260 266 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 267 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 268 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 269 και ΙΜΚΟ 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 269 και ΙΜΚΟ 26. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνονται. 270 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλη 13 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έμπλη 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έμπλη 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 282 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση 282. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ξεκάθαρα. 283, 284, έμπλη 16 και ΙΜΚΟ 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 285. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 286. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 287. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 297, 298, έμπλη 17, ΙΜΚΟ 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Μόνο η μισή ψηφίσατε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 2,99 και 300 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 307 και ΙΜΚΟ 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 308 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 313. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πηγαίνουμε στην 322. Υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την 322. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 323 παρα, ε, καταπίπτει. Ίμκο 39 επίσης. 326 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 328 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 327 ΙΜΚΟ 41 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Επιθυμείτε ηλεκτρονική επαλήθευση για το πρώτο τμήμα της 327 ε, και ΙΜΚΟ 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 329. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 330. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 331. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 332 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 333 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 334 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 334. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Εγκρίνεται. 340 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 336 υπέρ. Κατά. Αποχές θεωρώ πως εγκρίνεται αλλά δεν είμαι σίγουρος ηλεκτρονική επαλήθευση. Γιατί είναι 336. Πέρας. Εγκρίνεται. 341. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. 376 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 377. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές ηλεκτρονική επαλήθευση για την 377. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 378 έχει αποσυρθεί. 379 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. 33. Όλες αυτές καταπίπτουν. Συνεχίζουμε. Εγώ είμαι στη σελίδα 23. Συμβιβαστική 8. Τη βρήκατε? Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πήδαμε τις σελίδες. Πάμε στον Ρίχαρτ Τζέμπερ. 428. Υπέρ. Η κατά. Ο Ρίχαρτ Τζέμπερ θέλει ηλεκτρονική επαλήθευση. 426 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 427 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 425 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 429, 430 και ΙΜΚΟ 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 431 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονική επαλήθευση 431. Ψηφίσατε. Πέρας. Απορρίπτεται. 432 μέχρι ΙΜΚΟ 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνατε. Ήμικο 58 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές η ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε. Και ο Κάρλ Σλούτερ. Μάλιστα. Πέρας. Υπερεγκρίνεται. Ήμικο 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 435 καταπίπτει. Περνάμε λοιπόν στην 439. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 440. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 441. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 62. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4-4-2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση 442. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 443 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 444 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήμκο 63 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 446-447 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 445 καταπίπτει 448 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 450 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονική επαλήθευση για την 450. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Ίμκο 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 451. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ναι, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 4.52 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 481 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 10 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 492-493 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτονται. Συμβιβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 508. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 509 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 526 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 527 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σαφώς. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 528 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 529. Καταπίπτει 530 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 531 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 και 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5.35. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5.37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5.38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλη 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ενοποιημένη 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συνεχίζουμε με την 541 και ΙΜΚΟ 79. Υπέρ. Επαναλαμβάνω. Πρέπει να ψηφίσουμε την 541 και την ΙΜΚΟ 79. Τις βρήκατε? Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 544. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5.45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5.46 ΙΜΚΟ 80 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5.47, 5.48, 5.49 και ΙΜΚΟ 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Είμκο 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 550-51 Είμκο 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει 552 και πάμε 555 υπέρ. Dagegen κατά αποχές εγκρίνεται. Άλμα 599 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 600 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 602 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 603 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 604 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 605 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 606 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 607 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ζητάτε να ελέγξουμε την εμ 95. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Πέρας. Εγκρίνεται. Είναι 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 608 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 82 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ας την ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι για την 82. Πέρασε. Να εγκρίνεται. 36-31. Η 610 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 611 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 613 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 615 είπε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 616 Π. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88, 617 μαζί. ειπε Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 619 619-π Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 620 620-π Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η 90 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ενοποιημένη 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται Ήμικο 102 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμικο 103 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 104 ήμικο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 105 ήμικο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 629 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμικο 107 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 630 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Είμαστε στην 630. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε μια αρμονία, άλλο πράγμα. 60 υπέρ, 7 κατά. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 108 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 654 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6.33 6.34 μέχρι και 66 είναι μια ολόκληρη σειρά όλα αυτά μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται έμπλη 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 667 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 679 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 680 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 681 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 682 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 683 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 684 μέχρι 695 on μαζί όλες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 696 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 697 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε την 697 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. τα. 698 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 699 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 700 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 701 υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. 704 υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 710. Ρεμπέκα Τέιλορ υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 739 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφέ ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ την 739. Ψηφίσατε όλοι. Λείπουν 4, 3, 2, 1, τέλος. Εγκρίνεται. 740 επέ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Ήμικο 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 741 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 742 υπέρ. Α, καταπίπτει. Α, ψηφίζουμε την 109 τότε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα. 747 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 748 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 749 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 750 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 751 Μέχρι και 54 δεν ψηφίζονται. Ε, τα 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν κατάλαβα. Ηλεκτρονικά λοιπόν την 752. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 755 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλη 23 υπέρ κατά αποχές απορρίφθεται 756 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος γιατί δεν καταλαβαίνω από εδώ τι ψηφίζετε ψηφίσατε όλοι πέρασε εγκρίνεται 758 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ενοποιημένη 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 759 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 760 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 761 και ήμικο 130 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 763 και 767 μαζί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. ήμικο. 131 και η ΙΜΚΟ 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται η επόμενη καταπίπτει έμπληκος 4 υπέρ όχι και αυτή καταπίπτει α και αυτή τότε που πάμε τώρα 762. Ψηφιπέ. 762. Ξανά. Μου λένε ότι πρέπει να ψηφίσουμε την 762 γιατί τα προηγούμενα έχουν καταπέσει όλοι. Είπε. κατά, άποχες, εγκρίνεται. 769 είπε. κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έμπλη 27 είπε κατά αποχές απορρίπτεται. απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 770 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 771 μέχρι και 777 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Η επόμενη καταπίπτει και πάμε στην 779 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 780 και 797 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Apple 31 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ξέρω ψηφίζουμε τη 31 ηλεκτρονικά της Επιτροπής Απασχόλησης. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 34 υπέρ 28 κατά. Δεν κρίνεται λοιπόν. 782 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 783 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 784 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 785 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 786 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 33 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. 33 έμπλ. Ελέγχεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 787 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 788 μέχρι και 90 μαζί υπέρ. Οι ίδιες είναι κατά. Αποχές εγκρίνονται. 791 υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνονται. Ήμκο 134 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 794 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 795 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμικο 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα συνεχίζουμε με την τροπολογία 136 υπέρ κατά αποχές, δεν είναι σαφές. 136 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Φέρας. Απορρίπτεται. 138 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αμπλοκ τώρα. 839 μέχρι 844 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και άλλο μπλοκ τώρα. 137 μέχρι και 140 τη ΣΥΜΚΟ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 845 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 846 και ΙΜΚΟ 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 847 είπε Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 850 και 161 μαζί είπε Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Βάι Κέρπερ και Κράμερ 849. Ψηφιπέ κατά αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 849 ψηφίσατε όλοι λήξεις εγκρίνεται ΙΜΚΟ 2 και 159 ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε. Α, 160 θέλετε να την ελέγξουμε. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Απορρίπτεται. Έμπλ 3, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 848. Και οι τρεις επόμενες, υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικά καλύτερα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Εγκρίνονται. 8.53 μέχρι και 55 είπε. Κατά. Και αυτό θέλει ηλεκτρονικό έλεγχο του. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Εγκρίνεται. 8.56. Καταπίπτει. 140 και 8.57 μαζί. Είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8.59 είπε κατά άποχες εγκρίνεται έλεγχος έλεγχος 859 ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 860 και ΙΜΚΟ 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 861 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 862 π κατά άποχες απορρίπτεται 863 πέ κατά άποχες εγκρίνεται 864 πέ κατά αποχές απορρίπτεται 865 επέ κατά αποχές απορρίπτεται Ήμκο 145 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 866 καταπίπτει, όπως και οι επόμενες. Και πάμε στην 871 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε 871. Ψηφίσατε όλα πέρασα. Απέριφθη. 8,72 επέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8,73 επέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8,74 επέ. Κατά. Αποχές απορρίψεται. Ήμκο. 146 επέ κατά αποχές εγκρίνεται 875 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 876 μέχρι και 89 υπέρ κατά αποχές έλεγχος όλο αυτό το μπλοκ ηλεκτρονικά ψηφίζουμε ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 878 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 881 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 882 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μπλοκ. 883 μέχρι 887 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 890 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 892 πίπτη 895 υπέρ κατά αποχές πολλοί δεν ψηφίζουν ηλεκτρονικά λοιπόν την 895 ψηφίσατε όλοι Πέρα. Εγκρίνεται. Ήμκο 148 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 149 έμκο, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 150 έμκο, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 897 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 898 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 151 δεν καταπίπτει, την ψηφίζουμε είπε. κατά αποχές εγκρίνεται Σύμβασμος 26 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ 34 συγγνώμη 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 901 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 902 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 903 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ενοποιημένη 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλ 1 μέχρι και 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Οι δύο υπέρ. Κατά. Δεν ψηφίζεται. Ηλεκτρονικά λοιπόν ψηφίζουμε τη δύο. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 156 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 5 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 157 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 158 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικά. 158 τμήμα δεύτερον παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 163 ή 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. M6 κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 8 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 187 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 195 είπε, Κατά. Αποχές. 196 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 197 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 198 είπε κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ορίστε τρέχω πολύ 16 ηλεκτρονική απολύθευση. ψηφίσατε όλοι πέρας ε, σαφέστατα εγκρίνεται 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 207 ΙΜΚΟ 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 209 και 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.13 ειπε κατά αποχές εγκρίνεται 2.14 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται 2.15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΙΜΚΟ 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.16 είπε, κατά αποχές έλεγχος 2.16 ηλεκτρονική επαλήθευση Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.20 υπέρ. Κατά. Αποχές Έλεγχος για τη 2.20 ηλεκτρονικά. Δεν είμαι βέβαιος. Ψηφίσαμε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.21 υπέρ. Κατά. Αποχές. 2.21 ξανά παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην πρώτη τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα για την πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 52 υπέρ, 12 κατά με 3 αποχές. Και τώρα, τελική ψηφοφορία, η δεύτερη για το νομοθετικό ψήφισμα υπέρ. Ηλεκτρονικά διορθώνει ο Πρόεδρος, φυσικά. Ψηφίσατε όλοι. 52 υπέρ, 12 κατά και 3 αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Ντάγμαρ Ροτ Μπέρεντ. Και ευχαριστώ πολύ και τη γραμματεία, διότι γνωρίζω πόσο πολύ χρειάστηκαν για να επεξεργαστούν αυτόν τον κατάλογο και πώς επεξεργάστηκαν, πόσο σκληρή δουλειά έκαναν μαζί με τις ομάδες για να δημιουργηθεί αυτός ο κατάλογος. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν. Μισό λεπτό. Μη φύγετε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με την έκθεση του Πέτερ Εδώ έχουμε την ενοποιημένη τροπολογία 26. Υπέρ. υπέρ, κατά, αποχές, πολύ ωραία. Εγκρίνεται η ενοποιημένη 26, τροπολογία 111 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 13. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με την τροπολογία 12 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ.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 113 και ΙΜΚΟ 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ΙΜΚΟ 6 υπέρ. Κατά. Α, όχι, ήταν. Ε, την ψηφίσαμε αυτή, την ψηφίσαμε αυτή. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 117. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 116. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε ένα διάλειμμα μήπως. Μόνο πέντε ψηφίσατε. 116 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ήμκο 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρι... Α, απορρίπτεται. Ίνκο 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 118. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 119. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 120. Κατά τμήματα ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 120 ηλεκτρονική επαλήθευση στο δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ήμκο 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19. Υπέρ. Κατά. 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123 και ΙΜΚΟ 11 καταπίπτουν αυτές οι δύο. Συνεχίζουμε 124 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Λίμκο 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Unblock 22 και 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά. ηλεκτρονική επαλήθευση 131. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 132. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλε Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 133. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές η ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ήμκο 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 137. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 138 καταπίπτει. 29. Γιατί καταπίπτουν γιατί ψηφίστηκε η ΙΜΚΟ 17. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση 29. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Οι πράσινοι είχαν περισσότερες ψήφους. Ενοποιημένοι 4α. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένοι 4 β καταπίπτει. Σιγά σιγά προχωράμε στην 144 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 32 και 151 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 32 και 151. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ήμκο 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμικο 23. Καταπίπτει Ήμικο 23. Ίμκο 24 και Ίμκο 152. Εγκρίνονται 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154 και ΙΜΚΟ 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ παρακαλώ. Εγκρίνεται 155. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Συγγνώμη. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να ψηφίζετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Για δες, εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 135. Όχι 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ίνκο 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 161. 171. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 172. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 174. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 175. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 182. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 137. Υπέρ. Όχι, συγγνώμη. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38. Πώς είπατε? Ηλεκτρονική επαλήθευση στην 37. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38. Μάλιστα. Ξανά η ηλεκτρονική επαλήθευση. 38. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 183. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Unblock, ΙΜΚΟ 31 και ΙΜΚΟ 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. ΙΜΚΟ 31 και 32 ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με την 185 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη, κύριε Πρόεδρος. Ήμικο 33, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 189 και ΙΜΚΟ 35 τι είπατε κύριε Σλίτερ θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση ωραία ηλεκτρονικός έλεγχος ΙΜΚΟ 33 Ψηφίσατε όλοι. Μας λείπουν τέσσερις ψήφοι, τρεις πέρας εγκρίνεται. 189 και ήμικο 35 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 188 και ήμικο 34 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 208-209 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 20. μα όχι 2.19, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.20, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 228 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 230 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 232 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 233 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 2, 37 και 106 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 2, 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται ΕΜΠΛ 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται ενοποιημένη 27 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. 2.59 υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση 2.59. Ψηφίσατε όλοι. Χρησιμοποιήστε τα μηχανήματα παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι την 259. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.60 και 2.62 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται και αυτή, πιστεύω, αλλά ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 41. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Βιαστήκαμε. Από την αρχή. Η ηλεκτρονική επαλήθευση τροπολογία 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ήμκο 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 266. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση 266. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. Επιθυμείτε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Πράσινη και έλκ. Ορισμένοι το κατάλαβαν. 2,74 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2,75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2,76 υπέρ. Κατά. Απο... Απορρίπτεται. 3,43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμικο 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ήμικο 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 278 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές η ηλεκτρονική επαλήθευση 278. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 34, 34 υπέρ 31 κατά Εγκρίνεται. 45. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει το δεύτερο τμήμα. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 283 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 και 285 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 και 25 μπλοκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 286 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 28 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Ενοποιημένη 28. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Ήμκο 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.98. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Ήμκο 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 266 υπέρ. 299 με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 300 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 301 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 303 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 304 και ήμκο 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 62 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλη 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ίνκο 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.31. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.32. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3.33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3.34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3.35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3.36 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.38 υπέρ κατά αποχές ε, δεν είναι σαφές η ηλεκτρονική επαλήθευση 338 ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 3.40 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 3.42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ενοποιημένη 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3.45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3.46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62. Υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 62. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με την 347 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64. Υπέρ. Καλύτερα ηλεκτρονικός έλεγχος 348. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 35 υπέρ, 31 κατά. 50, 65 υπέρ, κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 64. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 3.49 υπέρ. Κατά. Καταπίπτει, φυσικά. Ήμκο 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 350. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 351. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 352. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 353. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλη 15. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 355. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 356 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 357 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. 357 η ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 358 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήμκο 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 359 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 382 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 385 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 και 69 unblock υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 386 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 387 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 80 πίπτη 388 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 389 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 81 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 82, πρώτο τμήμα. Σε δύο τμήματα ψηφίζουμε. Ήμκο 82, δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 83, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 390, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 391. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 392. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 393. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 394. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.96 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.97 υπέρ. Κατά. Αποχές Ηλεκτρονική επαλήθευση 397. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. εγκρίνεται. Αν σας ενοχλούμε την ώρα που τηλεφωνείτε, να διακόψουμε τη συνεδρίαση. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.98 και 3.99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΙΜΚΟ 85, ΙΜΚΟ 86, ΙΜΚΟ 87 και ΙΜΚΟ 88 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. ΙΜΚΟ 89 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 90 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 91 υπέρ. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλη 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλη 2 κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85. Καταπίπτει. Έμπλη 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλη 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλη 7. Υπέρ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 57 υπέρ, καμία κατά, 8 αποχές. Περνάμε στην δεύτερη τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 57 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, 7 αποχές. Συγχαρητήρια. Πέτερ Λίζε. Και πάλι ε, χίλια ευχαριστώ στην ώρα από τη γραμματεία. Εγώ ξέρω τι τράβηξε, πόσες ώρες και ε, πόσες μέρες χρειάστηκε. Άξιζε τον κόπο που την αναβάλαμε και πάει τώρα στην Ολομέλεια αυτή η ψηφοφορία, αυτή η έκθεση. Καλώς. Ε, Αγαπητέ Πέτερ Λίζε, πού πας. Λίζε θα προχωρήσουμε χωρίς εσένα. Κάτσε κάτω. Θέλεις εντολή. Ε, πρόεδρε, όπως και στην έκθεση Ροτ Parent, στην Ολομέλεια θα κάνουμε την τελική ψηφοφορία, διαβελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την έκθεση. Ευχαριστώ για την υποστήριξη και τους συνεργάτες της Γραμματείας που εργάστηκαν πράγματι πάρα πολύ σκληρά. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Η Ντάκμα Ροτ θέλει και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν πολύ σκληρή δουλειά, όντως. Καθόλου εύκολη για κανέναν από εμά. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους σκιώδης ηγητές. Κάναμε πολύ δρόμο μέχρι εδώ. Γνωρίζω ότι μέχρι την Ολομέλεια θα πρέπει να συνεργαστούμε και ελπίζω να το πράξουμε. Προσπάθησα στις συμβιβαστικές τροπολογίες να κάνω το τμήμα που μου αναλογεί και θέλω επίσης να πω ότι δεν ζητώ τώρα εντολή ε, να ψηφίσουμε πρώτα στην Ολομέλεια και μετά να αρχίσουν οι διαβουλεύσεις, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ταγμαρότη Πέρεντ και όλους σας που συμμετείχατε στην προσπάθεια αυτή. So, Και βεβαίως εδώ συμπεριλαμβάνονται και οι ε, υπάλληλοι των πολιτικών ομάδων για τις διαπραγματεύσεις. Χρειάζεται και αυτό το χρόνο του. Also vielen Dank Και πάλι ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους βοηθούς, τις πολιτικές ομάδες ε, και τους υπαλλήλους των πολιτικών ομάδων που έφτισαν αίμα για να γίνει έτσι ο κατάλογος ψηφοφορίας. Δεν τα κάνω μόνος μου εδώ. Καμιά φορά μπορεί να φαίνεται εύκολο. Οι υπάλληλοι των πολιτικών ομάδων μαζί με τη γραμματεία κάθονται με τις ώρες. Καλώς. Συνεχίζουμε όμως. Έχουμε και άλλα θέματα. 13. Και εδώ εισηγητής ο συνάδελφος ο Ρώση και ψηφίζουμε την τροπολογία 101. Ψηφιπέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 102 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 103 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 104 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 105 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 108 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107. Τσεκ. Ωραία. 108 ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. κρίνεται. 107 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική υπαριθμόν 1 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115 ειπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 117 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 118 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η ενοποιημένη 2 είπε. Κατά αποχές ξαναψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την ενοποιημένη 2 παρακαλώ ψηφίσατε όλοι Η Abstimmung ist jetzt geschlossen. πέρας 42 υπέρ 17 κατά σαφέστατα εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 dafür. 131 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ, κατά αποχές δεν είναι σαφές αυτό χρειάζεται έλεγχο 132 ηλεκτρονικό ψηφίσατε όλοι Πέρας. εγκρίνεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 135 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. πίπτη 136 και 137 είπε, Κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται.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 148 είπε. κατά, αποχές εγκρίνεται. 149 είπε κατά, αποχές εγκρίνεται. 151 είπε, κατά, αποχές εγκρίνεται. 150 είπε. κατά, αποχές εγκρίνεται. 152 είπε, κατά, αποχές απορρίπτεται. 153 είπε κατά, αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 3 είπε κατά αποχές ηλεκτρονικά. Λοιπόν, ελέγχουμε την ενοποιημένη τρία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. 159 λοιπόν υπέρ κατά απόχες δεν είναι σαφές ηλεκτρονικά και πάλι ψηφίζουμε την 159 ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 160 Επέ. κατά αποχές εγκρίνεται 161 Επέ. κατά αποχές εγκρίνεται 162 Επέ. κατά αποχές εγκρίνεται. 165 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. 166 τώρα είπε. κατά αποχές εγκρίνεται. 167 είπε. κατά αποχές εγκρίνεται. 168 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 172 επε κατά αποχές εγκρίνεται τώρα πού πάμε 173 Επέ. ορίστε για στιγμή να μου εξηγήσουν λίγο που πρέπει να πάω 174. μου λένε. είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 175 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 176 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 177 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 179 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 181 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 193 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 193. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίψετε. 194 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ κατά αποχές. Δεν είναι σαφές. Έλεγχος παρακαλώ 197. Ψηφίσατε όλα Πέρας. Απορρίπτεται. Η ενοποιημένη 4 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 202 καταπίπτει αυτή ποια θα πρέπει να ψηφίσουμε τώρα. 199 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα καταπίπτουν οι επόμενες και πάμε στη 204 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 205 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ. Απορρίπτεται. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές τώρα. Ελέγχουμε τη 211 ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ε, απορρίπτεται. Η ενοποιημένη, η συμβαστική συγγνωμή 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 2.18 υπέρ κατά αποχές απορρίφθεται 2.19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα 28 υπέρ κατά αποχές απορρίψεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίψεται 2.30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Mhm. Ich gebe einmal zu Protokoll. Wir haben gerade zwei. Τη 232 κατά λάθο την ψηφίσαμε, δεν έπρεπε. Δεν οφείλαμε ή δεν κάνει, εν πάση περιπτώσει, γιατί έχουμε γκρίνει τη 230. Να γραφεί στα πρακτικά, κάναμε αυτό το λαθάκι. Πάμε παρακάτω. 236 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 237 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 238 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψεται. Ενοποιημένη 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε με την τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6, 7, 6 υπέρ κατά αποχές 7 ειπε κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, τι να κάνουμε πέρασε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 Αποχέ εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 54 είπε κατά αποχές για να το ελέγξουμε αυτό 54 παρακαλώ ηλεκτρονικά ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται 55 ε, ε, είπε κατά αποχές εγκρίνεται 56 είπε κατά αποχές εγκρίνεται 57 είπε κατά αποχές εγκρίνεται 58 είπε κατά αποχές απερίφθη Α, όχι, ηλεκτρονικά ελέγχουμε την 58. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Μ, εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην προφορική τροπολογία. Παρθμόν 1 Είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 66 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 68 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 69 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 71 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 72 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 73 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 75 υπέρ, κατά 76 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται γιατί δεν ψηφίζουμε αν μπλοκ όλα αυτά τα πράγματα 86 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπε, κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέ, κατά αποχές έλεγχος για την 90 παρακαλώ ψηφίσατε όλοι Πέρας. 34 υπέρ, 25 κατά, εγκρίνεται. 92 υπέρ. Τι έγινε. Θέλετε να μπλοκ τις υπόλοιπες, 92 μέχρι και 100. Ε, ο εισηγητής τι έκανε, εν τη σοφία του με τους σκιώδεις, γιατί δεν το κανόνισε. Ε, ένα κατάλογο ψηφοφορίας έτσι. Λοιπόν, 92 μέχρι και 100 μαζί όλες υπέ κατά, αποχές, εγκρίνεται το σύνολο. Τελική ψηφοφορία και ηλεκτρονικά παρακαλώ αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ορίστε. Ομόφωνα. Ομόφωνα. 58. Άριστα πήρατε. Είναι όλοι ικανοποιημένοι. Μπράβο σα, κύριε Ορέστη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ του και οδησιακητέ και όλου του συναδέλφου που συνεργάστηκαν 100% και βεβαίω και στι υπηρεσίε μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ συμφωνώ και επαυξάνω τα συγχαρητήρια. Έχουμε και άλλη. Είναι τη συναδέλφου Κάτενμπαχ. Μέχρι 6,5 χρόνο έχουμε, μην ανησυχείτε, να ψηφίζουμε. Λοιπόν, είμαστε όλοι έτοιμοι με κάρτες και λίστες και όλα αυτά. Πάμε. Ρέγγι 2, ψήφι πέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 1, υπέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21, υπέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22, υπέ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 22 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. 27-24. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέγγι 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλη 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Τσεκ θέλετε. Έμπλ end. Ό,τι πείτε εσείς. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 35 υπέρ, 18 κατά. Μεγάλη πλειοψηφία υπέρ. Λοιπόν, 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και άλλο τσεκ. 26 ορίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίψατε. 25 ψήφι περ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, είναι σαφές. 32, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. έμπλη 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλ 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλ 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εμπλέ, 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλ 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλ 12 υπέρ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 δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη 47 Αρχίζει τώρα ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Mm, ισοψηφία απορρίπτεται. Έμπλο 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλο 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπελε 9 και ρέγγι 11 μαζί και τις μου και μου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίψεται. 50 υπέρ κατά αποχές τώρα τι έγινε ξανά η 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε την 54 παρακαλώ Ψηφίσατε όλοι πέρας. απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές απορρίψετε 61 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε 62 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές δεν είναι καθόλου σαφές ελέγχουμε την 64 ηλεκτρονικά Ψηφίσατε όλοι. Και πέρας. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλη 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλη 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλη 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλη 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτει. Τέμπλ 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. έμπλ 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστικό πακέτο 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 80 τώρα ψηφίπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ. Τσεκ γιατί ρέγγι 5 γιατί δεν ήταν σαφές. Την 5 λοιπόν ψηφίζουμε της περιφερειακής. Όχι, σαφέστατα γίνεται δεκτή. Δεν, δεν ξέρω το αποτέλεσμα, αλλά βλέπω τις ενδείξεις σας. Ε, 45-6. 81 ναι. Είπε. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Αλλά ας το ελέγξουμε για καλό και για κακό. Το 81. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασα. 28-21 εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφέ, 84 την ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα, Εγκρίνεται. 83 επέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85 είπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 10 υπέ Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ρέγγι 10 ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. Ρέγγι 6 ψηφίπε κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε 87 είπε. κατά δεν είναι καθόλου σαφές διότι τρεις φιλελεύθεροι σταμάτησαν να ψηφίζουν Την 87 λοιπόν την ελέγχουμε και πάλι. Ηλεκτρονικά. 87. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Α, ορίστε, εγκρίθηκε. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ρέγγι 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ρέγγι 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται οι δύο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 5 υπέρ κατά αποχές Θα την ελέγξουμε λίγο την 5 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίψετε. Η 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψετε 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ. Κατά. αποχέ απορρίπτεται. Η 9 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπρι, ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Έμπλε ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όλες μαζί τώρα 20 μέχρι και ένα πόπο όλες αυτές <laughs> μαζί την 20 και την 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται έμπλ β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλ σε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ, εδώ τι λέει τώρα, ε, αιτιολογική αναφορά ένα. Όχι, δύο. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπλ, αιτιολογική αναφορά τρία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και επόμενη τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ουφ, τελειώσαμε και με αυτό, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τελική. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 47 υπέρ, 3 κατά. Καμία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Κάντενμπαχ. So, Stunden 20 Minuten. Λοιπόν, 2 ώρες και 20 λεπτά, καλά είναι. Μπράβο σας που κρατήσατε και αντέξατε τόση ώρα ψηφίζατε, εργαστήκατε σκληρά και τώρα πάμε στο επόμενο θέμα στη Μέση διάταξη 15. Να περιμένουμε ένα λεπτό. Όσοι θέλετε να παραμείνετε, μην διστάσετε και όσοι θέλετε να φύγετε στο καλό. Σε ένα λεπτό συνεχίζουμε. So, ich Πιστεύω πως τώρα όλοι οι συνάδελφοι έχουν τη δυνατότητα ή να καταλήψουν την αίθουσα ή να καθίσουν πάντως όπως και να έχει κάντε σας παρακαλώ ησυχία διότι έχουμε και συνέχεια. Έχουμε τις τεχνικές εξόρυξης με χρήση και κιανιδίων, ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μπάνκι ζήτησε να γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Θα ζητήσω όμως πρώτα από την Κομισιόν να αρχίσει και παρακαλώ όσοι θέλετε να συμμετέχετε στη συζήτηση σηκώστε το χέρι. Η Κομισιόν έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι επικεφαλής της ομάδας ανακύκλωσης αποβλήτων και το Διευθυντηρίου για τα περιβαλλοντικά θέματα που ασχολείται με τα θέματα του Κιάνιου. Ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που προσκάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετάσχει και να συζητήσει για το θέμα του Κιάνιου και των ε, συστατικών του την εξόρυξη μετάλλων. Το θέμα είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο, διότι πρόσφατα υπήρξε ένα μείζον ατύχημα στην Παγιανμάρε. Το θέμα με το κιάνιο είναι ότι μόλυνε τους υδροφόρους ορίζοντες μετά από το ατύχημα αυτό και κάποια κράτη-μέλη ενέκριναν εθνικά προγράμματα για την απαγόρευση του κιανίου στην εξόρυξη μετάλλων. Το 2010 το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα για την απαγόρευση της χρήσης και ανιδίων στην τεχνική εξόρυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συζήτηση αυτή είναι πολύ έντονη ακόμη και σήμερα διότι υπάρχουν νέες εξορυκτικές ε, εγκαταστάσεις και εργοστάσια ε, νέα, νέες μάλλον νέες τεχνικές με τη χρήση των κιανιδίων σε πολλά κράτη-μέλη. Για να δούμε συνολικά την εικόνα, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι σε, πολλές, σε πολλά ορυχεία χρησιμοποιούνται, χρησιμοποιούνται τα κιανίδια ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στη Φινλανδία, τη Σουηδία. Νομίζω ότι υπάρχει ένα μικρό εργοστάσιο που χρησιμοποιεί αυτή την τεχνική και στην Ισπανία. Ε, πρόσφατα εκπονήθηκε μελέτη το 2010, η οποία αναφέρει ότι οι εναλλακτικές τεχνικές, ε, εναλλακτικές προς το ωκεάνιο στις εξορυκτικές βιομηχανίες δεν είναι βιώσιμες οικονομικά και έχουν παρόμοιους κινδύνους για το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι η τον των κιανιδίων από την εξωτερική βιομηχανία δεν ε, θα επιτρέψει να λειτουργήσουν χρυσορυχεία που υπάρχουν ακόμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ιδάλλως θα πρέπει να εξάγουμε τον χρυσό σε τρίτες χώρες για να γίνεται εκεί η επεξεργασία. Αρκεί να υπάρχουν όμως και εκεί αυστηροί κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει την ε, τοποθέτησή της για το θέμα της χρήσης και ανιδίων στη χρυσορυχία, στα χρυσορυχία μάλλον. Ε, Έχουμε πολλές συστάσεις για το θέμα αυτό. Είχαμε ανταλλαγές με συνεργάτες των και ευρωβουλευτές. Όμως να επιστήσω την προσοχή σας στο εξή. Η δήλωση του Επιτρόπου Ποτότσνικ στην συζήτηση στην Ολομέλεια από τον Απρίλιο του 2011. Στη δήλωση του επιτρόπου Ποτότσνικ έλεγε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα, συνο... ένα πλήρες σύνολο με πολύ αυστηρές απαιτήσεις για τις ε, τεχνικές εξόριξεις. Υπάρχουν διατάξεις για την, και στην οδηγία για τη μελέτη αντικτύπου της των μετάλλων καθώς και σε ε, μελέτες περιβαλλοντικές καθώς και στις οδηγίες για την περιβαλλοντική ευθύνη. Υπάρχει όμως και ένα συγκεκριμένο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται στη διαχείριση των αποβλήτων της εξωτερική βιομηχανίας. Η σχετική οδηγία προβλέπει πολύ αυστηρά όρια για τις συγκεντρώσεις ε, και ανιδίων στις διαδικασίες εξόριξης. Αυτές οι οριακές τιμές είναι πολύ αυστηρές και για να σας δώσω ένα συγκεκριμένο χειροπιαστό αποτέλεσμα για νέες εξορρυκτικές εγκαταστάσεις, η μέγιστη συγκέντρωση και ανεδίου που επιτρέπεται, βάσει της οδηγίας για τα εξορρυκτικά πόβλητα, είναι 200 φορές χαμηλότερη από ότι οι συγκεντρώσεις που απαντήθηκαν στο ατύχημα του Μπαγιαν πέραν αυτών των αυστηρότατων οριακών τιμών, τα περισσότερα χρυσορυχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναπτύξει ή τέλος πάντων θα πρέπει να προβλέψουν τεχνικές και διαδικασίες για την απομάκρυνση και την ε, ε, διάθεση του κιανιδίου προτού ε, διαθέσουν στο περιβάλλον τα απόβλητα της εξορρυκτικής διαδικασίας προκειμένου να περιοριστεί ο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ο Επίτροπος Ποτότσνικ επίσης είχε αναφέρει στη δήλωση του τότε στην Ολομέλεια, από τον Απρίλιο του 2011, ότι το να έχουμε την πλήρη εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου θα πρέπει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Στον τομέα αυτό έχουν γίνει πολλά έκτοτε. Πέρυσι, τα κράτη-μέλη εκπώνησαν εθνικούς καταλόγους για εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις εξόρυξης ή που έχουν πάψει τη λειτουργία τους, επειδή είχαμε ευρωπαϊκές κατευθυντήρες γραμμές για την επιθεώρηση των εξορυκτικών ε, εγκαταστάσεων που θα έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος της χρονιάς και αυτή τη στιγμή ξεκινούμε τη διαδικασία αναθεώρησης της εξορυκτικής των εξορρυκτικών τεχνικών που θα ορίσουν και το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, οι περιπτώσεις χρήσης και ανιδίων. Για τα χρυσορυχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει και προγράμματα τα οποία έχουν προσελκύσει μεγάλη προσοχή, όπως ε, η περίπτωση της Ρόζα Μοντάνα στην ε, Ρουμανία και αντιστοίχω και στην Ισπανία. Επιτρέψτε μου μια τελευταία παρατήρηση. Η συζήτηση για τα κιανίδια και τα, τις ενώσεις κιανιδιών δείχνουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια εξορθολογισμού των πόρων. Η ανακύκλωση είναι η ασφαλέστερη και η καλύτερη επιλογή για να ε, συνεχιστεί η εξόριξη χρυσού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ο χρυσός ε, και τα απόβλητά του δεν ε, προσωμιάζει με τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Κάτι που το, κάνει, το καθιστά ξεκάθαρο και η σχετική οδηγία. Και βεβαίως γι' αυτό θα υπάρξει και μια αναδιατύπωση της οδηγίας σύντομα. Ε, ωστόσο, για την ανακύκλωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι μπορεί να αντικαταστήσει την έλλειψη πρωτογενών υλών εδώ οι πρώτες ύλες πρέπει να προστατευθούν και με, βέβαια με την ανακύκλωση δεν θα φτάσουμε να καλύπτουμε 100% των αναγκών μας. Θα πρέπει να υπάρξει διασύνδεση μεταξύ του ποσού χρυσού που πρέπει να παράγεται και χρειάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1% της παγκόσμιας παραγωγής και της ζήτησης που υπάρχει για χρυσό από πολλές διαφορετικές, ε, από πολλούς διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να αυξήσουμε τα ποσοστά συλλογής και ανακύκλωσης με την πρωτογενή εξόριξη και να έχουμε και τέτοιους κανόνες που να διασφαλίζουν ότι οι εξορρεκτικές δραστηριότητες γίνονται με τρόπο που είναι ασφαλής και φιλικός για το περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι με το ισχύο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαιτέρως μέσω της οδηγίας για τα εξορρυκτικά απόβλητα, μπορούμε να επιδιώξουμε και να πετύχουμε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπάνκι ζήτησε το λόγο, ο κύριος Ματιά, κύριε κυρία Αντωνέσκου και η κυρία Χάση. Κύριε Μπάνκι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσίασε το θέμα, αλλά έχω πολλές απορίες και ήθελα να τις ε, αναφέρω. Επιτέλου έφτασε η στιγμή που η Επιτροπή Περιβάλλοντος ασχολείται με αυτό το τόσο σημαντικό θέμα, διότι συνειδητοποιώ ότι παρόλο που στις 5 Μαΐου 2010 ελήφθηκε με μεγάλη πλειοψηφία απόφαση να απαγορευτεί στα κρατημέλη η χρήση κυανιδίων στις εξορρυκτικές ε, τεχνικές, παρά την απόφαση αυτή στα τέλη του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπέβαλε πρόταση στο, ευρωπαϊκό Ευρωκοινοβούλιο όπως θα έπρεπε να είχε κάνει. Η απόφαση όμως αυτή είχε μεγάλη πολιτική σημασία. Οπότε δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την αδράνεια και την απάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, κυρίως γιατί ο Επίτροπος Ποτότσνικ και οι συνάδελφοι του συμφώνησαν ότι είναι πολύ πολλές οι εξορρυκτικές εγκαταστάσεις όχι μόνο τη Ρόζια Μοντάνα στη Ρουμανία, αλλά και σε άλλα κρατημέλη δεν πληρούν τα μέτρα ασφαλεία. Να δώσω και κάποια αριθμητικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τη Ρόζια Μοντάνα στη Ρουμανία. Και ήθελα κυρίως να με ακούσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για τα θέματα αυτά. Μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσει στην Ευρώπη για την επεξεργασία και την εξόρυξη χρυσού και ασημιού. Από το 2006 Έως το 2017 προβλέπεται να διαρκέσει η εξόριξη αυτών των μετάλλων στη Ρόζια Μοντάνα και επί 17 χρόνια εξορίσονται 42 τόνοι ετησίως στα 180 μέτρα βάθος όπου εκεί μπορεί να προκύψουν και περιβαλλοντικές καταστροφές. Ε, η περιοχή κατοικείται. Υπάρχουν κοντινά προστατευόμενες ε, περιοχές. Και να μην ξεχνάμε εδώ την φυσική καταστροφή του 2000, όπου η μόλυνση έπληξε πολύ μεγάλες εκτάσεις. Εξαπλώθηκε σε μεγάλες εκτάσεις. Δεν υπάρχει λοιπόν επαρκής προστασία αυτή της περιοχής, ούτε καμία εγγύηση ότι σε περίπτωση φυσικών έκτακτων ε, περιστατικών ε, με ένα σεισμό ή κάτι ανάλογο δεν θα προκύψει μια καταστροφή. Αυτό το θέμα δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο τη Ρουμανία αλλά και άλλες χώρες όπως συνέβη επί παραδείγματι με την μόλυνση ε, του 2000 βλέπουμε να υπάρχουν ε, φοβερές πιέσεις ε, το πολιτικό σκηνικό της Ρουμανίας, ασκούνται πιέσεις και προς τον κυβερνητικό συνασπισμό και υπάρχουν και μεγάλες αντιστάσεις προς τις εξορρυκτικές αυτές ε, δραστηριότητες. Ελπίζουμε λοιπόν ότι όταν υποβληθεί η πρόταση νομοσχεδίου από την πλευρά της ρουμανικής κυβέρνησης να ε, ασχοληθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το θέμα αυτό για να δει αν συνάδει με τον ε, δίκαιο της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, παρουσίασε τα στοιχεία της. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν θεωρεί ότι το προγραμματιζόμενο νομοσχέδιο της Ρουμανίας συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο. Αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό και από πολιτική άποψη. Επιπλέον, σήμερα, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει λάβει γνώση όλων των απαραίτητων στοιχείων. Γιατί από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουμε λάβει μια πρόταση εντό τη προβλεπόμενη προθεσμία, τον Δεκέμβριο δηλαδή του 2011. Τι έκανε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθυστερήσει τόσο πολύ Είχαμε μια πλειοψηφία που ξεπερνούσε τι 200 ψήφου τον ε, Μάιο του 2011. Ήθελα λοιπόν να μα πει ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ή καλύτερα εάν ζήτησε από τις κυβερνήσεις των εν λόγω χωρών της Ουγγαρίας λόγου χάρη ε, έγγραφα που να καταγράφουν τις ζημιές ε, να προβλέπουν το τι θα γίνει σε περίπτωση που προκύψει ζημιά από τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές. Είναι σημαντικό αυτό το τι θα γίνει με τη χρήση των κυανιδίων στην εξόριξη χρυσού. Ε, ξέρουμε ότι η βουλγαρική κυβέρνηση λόγω χάρη αρνήθηκε την άδεια σε, της χρήσης των ε, ουσιών αυτών στην εξόριξη χρυσού και προβλέπει μια εναλλακτική μέθοδο Σε κάθε περίπτωση ηλεκτρονικά μέσα υπάρχουν. Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Και μεταξύ άλλων είναι πολλά τα απόβλητα από την εξόριξη χρυσού που θα μπορούσαν να ανακυκλώνονται. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε τέτοιες διατάξεις, τέτοιους κανόνες που να μπορέσουν να διευκολύνουν την λειτουργία των χρυσορυχείων. Λόγω χάρη στην ε, Σουηδία υπάρχει ένα χρυσορυχείο όπου τα δύο τρίτα της παραγωγής γίνεται με την ανάκτηση χρυσού μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί πολύ πιο σοβαρά υπόψη η τοποθέτηση του Ευρωκοινοβουλίου, διότι το Κοινοβούλιο Προσωπεί 550 εκατομμύρια πολίτε. Είμαστε το μεγαλύτερο εκλεγμένο κοινοβούλιο παγκοσμίω. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα λαμβάνει λιγότερο, περισσότερο σοβαρά υπόψη. Ε, δεν μπορεί να είναι παραδεκτό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τέτοιε αποφάσει του Ευρωκοινοβουλίου αποκοιμιέται. Σήμερα, μετά από μια τέτοια ανταλλαγή απόψεων, ε, θα πρέπει ένα τόσο σημαντικό θέμα να το ε, εξετάσουμε πολύ σοβαρά σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Επιτροπή Περιβάλλοντο του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστούμε, κύριο Γκερμπάντη. Ο κύριο Σταμπάντη, μάλλον. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριο Ταμπάντη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με τον ε, συνάδελφο και ευχαριστώ για την πρωτοβουλία οργάνωσης αυτής της συζήτησης. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα, με ένα θέμα πολύ σοβαρό που αφορά ε, τις σχέσεις Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί χρόνια έχει παραμείνει απαθής. Το Ευρωκοινοβούλιο από το 2010 έχει εγκρίνει απόφαση ε, και εγώ ήμουν ένας από τους συνεισηγητές για το ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά τα δύο τρίτα, με τα δύο τρίτα της... Ε, ε, με πλειοψηφία δύο τρίτων στο Κοινοβούλιο. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν προσωπικά τον πρόεδρο της Επιτροπής του Περιβάλλοντος. Δεν θα έπρεπε να απευθύνουμε μια επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο ε, ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξουμε μεγάλη προσοχή το θέμα τη Ρουμανίας. Υπάρχουν τρία σημεία που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραβλέψουμε. Οι τεχνικέ εξο... με χρήση και ανιδίων προβλέπουν πολλέ διαφορετικέ εναλλακτικέ. Γιατί η ρουμανική κυβέρνηση δεν ζητά από τους επενδυτές να προτείνουν ε, επιλογή μεταξύ των διαφορών αυτών εναλλακτικών που χρησιμοποιούνται ήδη στη Σουηδία και τη Φιλανδία και θα προσέφεραν μεγαλύτερα επίπεδα προστασία σε σχέση με τι τεχνικέ που ε, αυτή τη στιγμή πρόκειται για οικονομικού και μονολόγου να εφαρμόσει η Ρουμανία. Γιατί δεν χρησιμοποιείται μια τεχνολογία κυκλιστού κυκλώματο που θα ήταν πολύ ασφαλέστερη και για το περιβάλλον αυτό. Θα πρέπει να επιβληθεί στου επενδυτέ. Έπειτα, σε δεύτερη φάση, εμεί στην περίπτωση οποιασδήποτε φυσική καταστροφή δεν έχουμε καμία εγγύηση ότι θα μπορέσουν να αποκατασταθούν οι περιβαλλοντικές ζημιές που ίσω προκύψουν. Να θυμίσουμε την ε, περίπτωση της κόκκινη λάσπης και την καταστροφή αυτή ε, στην Ουγγαρία. Οι ζημιές ήταν τετραπλάσιες σε σχέση με ε, την, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρεία που προκάλεσε αυτό το ατύχημα. Ε, μην ξεχνάμε λοιπόν ότι μιλάμε για πολύ σοβαρέ απειλέ, πολύ σοβαρού κινδύνου. Γιατί το ρουμανικό κράτο, η κυβέρνηση δεν επιβάλλει στην εν λόγω επιχείρηση μια τέτοια υποχρέωση. Γιατί δεν επιβάλλει κάτι πιο δεσμευτικό. Ε, λόγου χάρη, είναι αστείο να ασχολείται κανείς με την ε, αποζημίωση 500 εκατομμυρίων ε, για τη χρήση των κιανιδίων σε σχέση με το τι καταστροφές μπορεί να προκύψουν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Δεν έχουμε τίποτε στα χέρια μας από αυτή την πλευρά. Δεν ξέρουμε ούτε καν ποιοι είναι ενδεχόμενοι κίνδυνοι. Γι' αυτό προτείνω αυτά τα τρία στοιχεία οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη και να μελετηθούν θα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο μιας κοινή απόκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ρουμανικής κυβέρνησης, τις ανησυχίες όλων μας. Διότι πραγματικά όχι μόνο η Ρουμανία θα πρέπει να ανησυχεί, αλλά και οι όμορες χώρες. Λοιπόν, ε, Πρόεδρε, επιμένω, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε πλέον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ε, επί ε, εξέταση του θέματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τις υπάρχουσες ε, διατάξεις και τα νομοθετικά μέτρα, αλλά να λάβει συγκεκριμένη πρόνοια, γιατί υπάρχουν εδώ σοβαροί παροδικοί κίνδυνοι. Ευχαριστώ. πολύ, κύριε Αντωνίασκου. mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță este un subiect foarte Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάμε για ένα θέμα πολύ σοβαρό. Ένα θέμα ε, που θα, πρέπει να, θα έπρεπε να έχει απασχολήσει ήδη την Επιτροπή μας και οπωσδήποτε πρέπει να συζητήσουμε. Υπάρχουν κάποιες ε, μεμονωμένες πρωτοβουλίες, ιδιωτικές πρωτοβουλίες που έχουν ε, δεχτεί πολλέ κριτικέ σε σχέση με το εγχείρημα τη Ρώσια Μοντάνα. Καταλαβαίνετε ότι για τη Ρουμανία ε, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα τη Ρώσια Μοντάνα. Έχει προκαλέσει μεγάλε κοινωνικέ εντάσει. Υπάρχουν σοβαρότατε αντιπαραθέσεις και σοβαρή αντίσταση από διαφορετικές πηγές. Είναι πολλοί αυτοί που αντιτίθενται σε αυτό το πρόγραμμα και πολιτικοί και απλοί πολίτες. Και σε ό,τι αφορά τη δική μας την Επιτροπή, νομίζω ότι πολλά ερωτηματικά παραμένουν αναπάντητα. Όχι μόνο προς τη χρήση ή τη μη χρήση και στις εξωτερικέ τεχνικές, αλλά ως προς τις διαστάσεις του ε, προγράμματος και τις υπόλοιπε τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη Ρόζα Μοντάνα. Το επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας που παράσχεται από τους ε, επενδυτέ είναι ένα αντικείμενο αμφιλεγόμενο η χρήση των βέλτιστων πρακτικών δεν υφίσταται καν σε αυτή την περίπτωση. Ε, και ως προς τα χρυσορυχεία, εδώ έχει, πάρει τελείως, ε, έχει περάσει σε τελείως δεύτερη μοίρα. Μιλάμε για την απομάκρυνση πολλών πολιτών, 370.000 θα πρέπει να ε, μετακινηθούν, 16 χωριά θα μετακινηθούν από τα 17, τα 3, θα πληγούν σοβαρότατα και το τοπίο στη Ρόζια Μοντάνα θα αλλάξει διαπαντός. Παρά τις ε, βεβαιώσεις των επενδυτών ότι θα προσπαθήσουν να μετριάσουν ε, τις ε, αλλαγές, οι ειδικοί λένε ότι και το περιβάλλον και το τοπίο θα αλλάξουν ανεπανόρθωτα. Γι' αυτό η συζήτηση αυτή πρέπει να ενσκύψει και στα θέματα του περιβάλλοντος, αλλά και του τι είδου ανάπτυξη θέλουμε να προωθήσουμε στην Ευρώπη. Δεν ε, θα απέκλεια από τη συζήτηση αυτή και το να ε, κοιτάξουμε τις ανάγκες για επενδύσεις. Σίγουρα πρέπει οι εξωτερική μας πόροι να εμπλουτιστούν και, να εμπλουτιστούν κι άλλο. Όμω αυτά όλα πρέπει να γίνουν με τρόπο που να μην παραβλέπει την αηφορία καθώς και την, ε, το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή αυτή πολλοί από τους οποίους είναι άνεργοι. Θα πρέπει λοιπόν όλα να τα βάλουμε στη ζυγαριά. Ε, υπάρχουν υπερβαλλοντικές ε, διατάξεις και απαιτήσει, ε, η υπερβαλλοντική προστασία, αυτό που ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ θέλω να σταθώ. Γιατί θα ήθελα να καταλάβουν οι συνάδελφοι ότι ο τρόπος με τον οποίο η ρουμανική κυβέρνηση επέλεξε να προωθήσει αυτό το εγχείρημα είναι με νομοσχέδιο. Το Ελήθη νομοθετική δράση. Η κυβέρνηση όμως δεν ανέλαβε πολιτική ευθύνη. Για πολιτικούς λόγους δεν θέλησαν να διακινδυνεύσουν το πολιτικό τους κεφάλαιο εκτιθέμενοι με αυτό το ε, εγχείρημα, διότι αντιτίθεται η κοινωνία των πολιτών σε, αυτήν την, ε, σε αυτό το εργοστάσιο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος βέβαια, μέρος της κυβέρνησης δηλαδή, δεν συγκατατέθηκε. Το Κοινοβούλιο πάντως εξέτασε προς έγκριση το νομοσχέδιο χωρίς να υπάρχει συγκατάθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ανεπάρκειες αυλεψίες και ε, ελλείψεις παρουσιάζει αυτό το πρόγραμμα. Το θέμα βεβαίω είναι όχι απλώ να αποδοθούν ευθύνε, αλλά το τι θα κάνει και το Υπουργείο Δικαιοσύνη που κλήθηκε να γνωμοδοτήσει. Εκεί το πόρισμα του Υπουργείου Δικαιοσύνη ήταν ένα πραγματικό κατηγορό. Είπε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι αντισυνταγματικό και προβλέπει άδειε εξόριξη για μια εικοσαετία, κάτι που είναι εντελώ παράνομο. Όλα αυτά θα έπρεπε να μα απασχολήσουν και να μα το θορυβήσουν. Πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και να τα σκεφτεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κατά την αποτίμηση του πώ έχουν τα πράγματα στη Ρώσια, Μοντάνα και τι γίνεται με αυτό το πρόγραμμα. Α είμαστε τέλο πάντων ειλικρινεί. Ο λόγο που οργανώθηκε αυτή η συζήτηση είναι ακριβώ αυτό. Η Ρώσα Μοντάνα και το εργοστάσιο, καθώ και οι πρόσφατε αντιπαραθέσει και διεξηφισμοί για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε, κυρία Σατουχάση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτω με του Ούγγρου ε, συναδελφού και συμμερίζομαι την απογοήτευσή τους ε, για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρακολούθησε αυτά που ζήτησε το Κοινοβούλιο πριν από μία τριετία, δηλαδή την απαγόρευση χρήσης και ανιδίων στις τεχνικές εξόριξεις. Θα ήθελα να θέσω τρία συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως ό,τι αφορά το πρόγραμμα της Ρωσία Μοντάνα. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει πραγματικά ότι χρησιμοποιούνται εκεί οι βέλτιστες τεχνικές εξόριξης. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για τα υπολείμματα είναι οι ασφαλέστερες. Να θυμίσω το τραγικό ατύχημα που είχαμε πριν λίγα μόλις χρόνια στην Ουγγαρία με την καταστροφή της κόκκινης λάσπης, όπως ε, έγινε γνωστή. Ένα από τα διδάγματα αυτού του περιστατικού ήταν ότι το εύστοχον των περιβαλλοντικών μελετών τύπου είναι κάτι σημαντικό. Ακόμα και οι δραστηριότητε όμως ε, παρακολούθησης και επιθεώρησης δεν ήταν επαρκής. Τι θα κάνει για αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περίπτωση της ε, Ρώσια Μοντάνα. πώ θα υπάρχει περιβαλλοντικό έλεγχος μεταξύ των οποίων και για, για τα υπολείμματα και την επεξεργασία τους. Και μετά κάποια σχόλια. Πρώτον, είναι μια πραγματική αντίφαση το να λέμε ότι θα χρησιμοποιώ τις καλύτερες τεχνικές εξόρυξης από τη μια και από την άλλη ε, μία τεχνική να προτιμάται σε σχέση με άλλες. Τα κιανίδια δηλαδή. Και η μόνη αιτιολόγηση είναι ότι περιορίζεται το κόστος. Ο περιορισμός του κόστους είναι ένα πράγμα και κάτι τελείως διαφορετικό η ε, καλύτερη τεχνική. Εάν οι εναλλακτικέ είναι λιγότερο ασφαλείς, αυτό είναι επιχείρημα, αλλά το κόστος είναι τελείως διαφορετικό. Εάν μια εναλλακτική τεχνική που δεν χρησιμοποιείται ευρέω είναι ασφαλέστερη από τη χρήση ανιδίων, αλλά σε κάποιο βαθμό πιο δαπανηρή, μπορεί όμως να περιοριστεί το κόστος της με εξορθολογισμό στη χρήση. Το ξέρουμε αυτό από την ιστορία των ε, περιβαλλοντικών υποθέσεων και καινοτομιών. Υπάρχει ένας μακροσκελής κατάλογος τέτοιων περιπτώσεων. Ε, δεν ε, ε, ικανοποιήθηκα με την επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί ως αιτιολόγηση μόνον το προ περιορισμένο κόστο για τη χρήση και στις στι τεχνικές. τεχνικέ. Έπειτα, το δεύτερο σχόλιο μου πιο συγκεκριμένα έχει να κάνει με, με το περιεχόμενο του κιανιδίου. Βάσει τη οδηγία των εξορρυκτικών αποβλήτων του Μαΐου της φετινής χρονιάς, το μέγιστο όριο συγκέντρωσης κιανιδίου στα νερά που παραμένουν ως απόβλητα είναι 25, της, είναι 25 μέρη ανά εκατομμύριο. Αυτό σημαίνει 25 ε, μιλιλίτρα στο ε, λίτρο. Η γραμματεία της Επιτροπής μας μας λέει ότι μιλάμε για 20 μικρογραμμάρια ανά λίτρο. Αυτό είναι το όριο εντός του τοπίου. Ε, πεθαίνουν τα ψάρια, αλλά και οποιοδήποτε άλλο είδος μπορεί να πεθάνει. Αυτό λοιπόν που επιτρέπεται για τα απόβλητα, τα νερά των αποβλήτων, είναι 100 φορές πιο δυνατό από αυτό που σκοτώνει τα ψάρια. Δεν ακούγεται και πολύ λογικό. Και το τρίτο μου σχόλιο. Χθες μόλις έμαθα ότι η Φινλανδία έχει χρησιμοποιηθεί από τον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας ως παράδειγμα στην, εξατρα... στην εκστρατεία του. Προσπάθησε να διαφημίσει τη χρήση και ανιδίων στι εξωτερικέ τεχνικές, χρησιμοποιώντας τη Φιλανδία ως παράδειγμα. Ο συνάδελφος, ο κύριος mm. συγγνώμη, μόλις έπαθα ένα κενό μνήμης. Τζάμπα, εσύ αναφέρθηκες στις τεχνικές κλειστού κυκλώματος στη Φινλανδία. Υπάρχει εξορρυκτική βιομηχανία, η καναδική Gabriel Resources, η οποία στην Πορκίτια, σε αυτήν την περιφέρεια, έχει κάνει εκστρατεία κατά του ψηφίσματος που ενέκρινε το Κοινοβούλιο πριν από μια τριετία. Λένε ότι η δική τους διαδικασία είναι μια διαδικασία κλειστού κυκλώματο, κάτι που δεν ισχύει. Διότι εκ των υστέρων είχαμε τουλάχιστον ένα περιστατικό όπου τα ανώτατα όρια συγκέντρωσης και ανιδίων στα νερά των αποβλήτων ε, ξεπεράστηκαν. Και τα απόβλητα αυτά ήταν ιδιαίτερα ογκώδη για, τις, ε, για, τα, νερά αυτά που χρησιμοποιούνται για, την, για τον καθαρισμό. Για τις δεξαμενές λένε οι υπεύθυνοι της εταιρείας ότι οι μετρήσεις που έγιναν εκεί δεν ήταν αρκετές για να μετρηθεί ο αντίκτυπος στους υδροφόρους ορίζοντες, τα εδάφη, για να υπολογιστεί ο κίνδυνος για τα ψάρια, κατά τα στοιχεία που διαθέτω, δεν Υπάρχουν ε, πληροφορίες για νεκρά ψάρια γύρω από το εργοστάσιο, αλλά υπάρχουν και τα νερά των ποταμών που ε, βρίσκονται κατά άντι του εργοστασίου. Λοιπόν, δεν συμφωνώ ότι η Φιλανδία είναι κανένα υπέροχο παράδειγμα της χρήσης και ανιδίων στις εξωτερικές τεχνικές, με τρόπο απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον και μάλιστα σε κάποια άλλα ορυχεία, Είχαμε σοβαρά ατυχήματα, όχι με τα κιανίδια, αλλά με φράγματα ή με δεξαμενές που ράγισαν. Με τις περιπτώσεις θείου και θείουχων αλάτων και άλλων βαρέων μετάλλων που εκχύθηκαν στο περιβάλλον. Είναι αρκετά σαφές για τους Φιλανδούς πάντως και την κοινή γνώμη στη χώρα μας ότι η μεταλλουργία είναι μια πολύ επικίνδυνη βιομηχανία. Ο Επίτροπος Ποτότσνικ έχει κάνει πολύ λόγο για, και με τρόπο θετικό μάλιστα έχει αναφερθεί στην ε, εξορθολογισμένη χρήση των πόρων. Εάν ήταν σοβαρός ως προς αυτό το θέμα, θα έπρεπε να πιέζει περισσότερο και να απαιτεί ανακύκλωση των ε, ηλεκτρονικών αποβλήτων λόγου χάρη. Ε, ένας τόνος ε, κινητών τηλεφώνων περιέχει 50 φορές περισσότερο χρυσό από ότι ε, τα απόβλητα των χρυσορυχείων ε, αυτή τη στιγμή. Θα ήταν πιο αποτελεσματικό να συγκεντρώναμε απόβλητα της ε, βιομηχανίας ηλεκτρονικών και θα περιορίζαμε και τα ορυχεία και τα χρυσορυχεία ανά την Ευρώπη. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τα αστικά απόβλητα, ώστε να έχουμε και κάποιο είδους αστική εξόρεξη, για να το πω έτσι. Αυτά ο Επίτροπος Ποτότσνικ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να τα προωθούν και να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Τούρκης. Tisztelt Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε. Είμαι ένας Ούγγρος της Ρουμανίας. Και ενδιαφέρουν και οι δύο χώρες το ίδιο, ως προς το ζήτημα μάλιστα που συζητάμε. Η ρήπανση ε, έχει, έπληξε το 2010 την Ουγγαρία κυρίως, αλλά και τη Ρουμανία. Η Ρώσια Μοντάνα και το όλο εγχείρημα θα μπορούσε να έχει σοβαρό αντίκτυπο και επιπτώσεις όχι μόνο στο ρουμανικό περιβάλλον, αλλά σε όλη την υδρογραφική λεκάνη του Μπίσκου. Δηλαδή και στις ε, όμορες περιοχές και χώρες. Να πω ότι πρόκειται για ένα θέμα που αφορά από κοινού ε, την ε, κεντρική Ευρώπη και την Ανατολική Ευρώπη συνολικά. Το λέω αυτό ε, εκφράζοντας την πλήρη μου αλληλεγγύη και προς τους Ούγκρους συναδέλφους και προς τις δεκάδες χιλιάδες πολιτών που ήδη από ένα μήνα περίπου διαμαρτύρονται στη Ρουμανία. Και εγώ συμμετείχα σε διαδήλωση στο Κλούζ όπου 10.000 νέοι διαμαρτυρήθηκαν, κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν. Και με μεγάλη αίσθηση ευθύνης τους ως πολίτες και με μεγάλη ευσυνειδησία ε, τάχθηκαν υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε το θεμελιώδες ζήτημα εδώ. Και ποιο είναι αυτό. Το εξής. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε με μια πλειοψηφία των δύο τρίτων θα έπρεπε να έχετε κάποιο πολιτικό βάρος. Ας μην παίζουμε με τη δημοκρατία, το είπε και ο κ. Μπάνκι. Εδώ εκπροσωπούμε 500 εκατομμύρια πολίτες. Εάν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η απόφασή μας είναι τόσο ασήμαντη μια απόφαση που είναι καθόλου ανόμιμη, ε, ας μην καθόμαστε καν να συζητάμε το όλο θέμα. Δεν έχει κανένα νόημα. Εγώ έχω επικρίνει επανειλημμένο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τον Επίτροπο Ποτότσνικ, διότι υποψιάζομαι ότι εδώ κάτι υποκρύπτεται για κάποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει δράσει κατά αυτόν τον τρόπο και έχει τις ευθύνες της που θα πρέπει να αναλάβει. Και στη Ρουμανία υπάρχουν όμως επιπλοκές και εκεί το, η δημοκρατία δεν λειτουργεί εύρυθμα. Ήδη στο από τον Αύγουστο η κατάσταση που επικρατεί είναι ε, τραγική και κομική ταυτόχρονα. Μιλάμε για μια σειρά νομοσχεδίων που έχουν κριθεί αντισυνταγματική. ο ένας υπουργός κατηγορεί τον πρόεδρο Μπασέσκου, ο πρόεδρος της συγκλήτου της Γερουσίας, συγγνώμη, κατηγορεί κάποιον άλλον ε, πολιτικό ηθήνοντα. Καθημερινά, λοιπόν, βγαίνουν στις ειδήσει χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ότι πρόκειται για νομοσχέδια αντισυνταγματικά. Πρόκειται για, μια, ε, για ένα μπραντεφέρ μεταξύ των ε, κομμάτων και αφορμή είναι ακριβώς αυτό το νομοσχέδιο. Εδώ μιλάμε για χειραγώγηση. Στο... Ο κύριος Πλούμ που είναι υπουργό. Είχε έρθει εδώ το 2010, ήταν μέλος του Ευρωκοινοβουλίου και ψήφισε μαζί μας κατά της τεχνικής εξόρυξης αυτής με τη χρήση και Και αυτή τη στιγμή έχει περάσει στην αντίπερα όχθη στο αντίπαλο στρατόπεδο. Ε, ο Επίτροπος Ποτότσνικ είχε πει και εδώ απλώς αναφέρω τα λόγια του, ότι ο ρουμανικός λαός, το μεγαλύτερο μέρος της ρουμανικής κοινή γνώμης, είναι υπέρ αυτών των τεχνικών εξόριξης. Μα θα πρέπει να καταλάβουμε, ε, ε, ε, συνάδελφοι, ότι ο σκεπτικισμός κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλο ένα και περισσότερο εξαπλώνεται. Η κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει οδηγήσει σε κρίση αξιοπιστίας κυρίως και εμπιστοσύνης. Ε, πιστέψτε με, στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία μειώνεται διαρκώς, όχι μόνο σε αυτές τις δύο χώρες προφανώς, αλλά και σε αυτές η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η συμπεριφορά, η παραγνώριση των ε, επιθυμιών των πολιτών δεν μπορεί να μας οδηγήσει πουθενά. Δείτε τι έγινε στην Ελλάδα. Σε αυτή την επιτροπή είχαμε οργανώσει την τελευταία μας συνεδρίαση και μια ακρόαση σχετικά. Είχαμε συζητήσει θέματα που αφορούν την Ισπανία. Ε, ακούσαμε τι γίνεται με τις διαμαρτυρίες εκεί. Βλέπουμε ποιες είναι ο αντίκτυπος του σχεδιασμού τέτοιων πολιτικών. Και μην ξεχνάμε και περιπτώσεις όπως αυτές και ατυχήματα όπως αυτά του Τσερνομπίλ και της Φουκουσίμα. Να επιμείνω λοιπόν εδώ. Υπήρξε πλειοψηφία 82% αυτού του, Ευρω... αυτού του Κοινοβουλίου υπέρ της συγκεκριμένης απόφασης. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα πρέπει να τηρήσει μια συγκεκριμένη στάση. Και απευθυνόμενοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφράσει τις δίκαιες ανησυχίες μας και τις απαιτήσει μας. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπουμε πολλούς νέους συναδέλφους τώρα, αλλά ε, θα ακούσουμε και μια συνάδελφο που ασχολείται εδώ και καιρό με το θέμα που είναι η κυρία Κρίστα Κλάς. Ευχαριστώ. Ε, ε μας ε, ξανάρχονται οι αναμνήσεις και το ξέρω πολύ καλά αυτό το θέμα της Ρόζα Μοντάνα. Όταν ήμουν ε, αρμόδια το 2006, εισηγήτρια για αυτό το θέμα για τα απόβλητα των ορυχείων. Πήγαμε στη Ροζία Μοντάνα και ε, υποσχεθήκαμε κάποια πράγματα στον κόσμο εκεί, δηλαδή Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα απόβλητα των ορυχείων και για τα κατάλληλα και ότι η Ρουμανία ως ευρωπαϊκή χώρα μετά θα πρέπει να τηρήσει την οδηγία αυτή. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτή την υπόσχεση και πάνω από έκπληκτη δηλώνω και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς μπορεί να έρχεται σήμερα εδώ και να δηλώνει ότι χρειαζόμαστε φυσικούς πόρους και μάλιστα ε, χρυσό. Και ποιος δεν θέλει χρυσό, ποιος δεν αγοράζει χρυσό. Ε, δεν τον απεμπολούμε έτσι το χρυσό, ούτε τον αφήνουμε να κείται μέσα στα ορυχεία. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολη ακριβώς ε, η θέση του χρυσού για να το βρει στη φύση σκάβουν ολόκληρα βουνά και ε, δεν ξέρω πώς ε, στη συνέχεια μπορούμε να αποτρέψουμε βλάβες στο περιβάλλον. Γιατί δεν επιτρέπεται επειδή θέλουμε χρυσό να δηλητηριάζουμε και το νερό, επειδή χρησιμοποιούμε τοξικές ουσίες για να βγάλουμε το χρυσό. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα κατάλοιπα των ορυχείων δεν είναι αυτές κατευθυντήριες γραμμές να μην ε, έχουμε περιβαλλοντικές ε, ε, καταστροφές, να επαναφέρουμε στην προηγούμενη κατάσταση το χώρο, να χωρούμε σε αποκατάσταση του περιβάλλοντος και της φύσης κτλ. Είναι πολύπλευρη αυτή η ιστορία και η ρουμανική κυβέρνηση πούλησε ε, την περιοχή αυτή και θέλει μια καναδική εταιρεία τώρα να κάνει την εξόριση. Δεν πάνε να είναι και καναδική εταιρεία. Πρέπει να τηρήσει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ε, αυτή η ιστορία στη Ροζίγια Μοντάνα ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις και τους όρους και τα προαπαιτούμενα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα κατάλοιπα και τα απόβλητα της εξορρεκτικής βιομηχανίας ερώτηση. Θέλω σαφέστατη απάντηση χωρίς ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς ως Κοινοβούλιο έχουμε δώσει το λόγο μας εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος, ο συναδελφός Σόγκο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι ένας από εκείνους που έστειλαν επιστολή στον Επίτροπο Η Φουκουσίμα και η καταστροφή στην Ιαπωνία δεν είναι, δεν είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο έχουμε και, και εμείς εδώ αρκετά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντιδρά. Περιμένει πρώτα να συμβεί κάποιο σκάνδαλο και μετά να αντιδράσει, όπως για παράδειγμα με την περίπτωση των ε, Ρωμά στη Γαλλία. στον... στο θέμα αυτό, στην εξορρυκτική βιομηχανία, τι περιμένετε, περιμένετε να γίνει κάποια καταστροφή, μια τεράστια καταστροφή πάλι. Ε, απαντήστε μας, σας, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ας ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ε, υπευλήθησαν πολλές ερωτήσεις, σας κατηγόρησαν και τώρα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε στα πάντα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, πιο σημαντική ερώτηση ίσως ήταν εκείνη του κυρίου Μπάνκι και του κυρίου Ταπάντζη. Οι καθυστερήσεις στη συμμόρφωση με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εξόριξη. Κατά την άποψή μας δεν έχει συμβεί καμία καθυστέρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε ξεκάθαρα την απόψή της για το θέμα αυτό. Προσπάθησα να το κάνω και σήμερα εγώ. Ο Επίτροπος Ποτόσνικ το έχει κάνει στο παρελθόν, γραπτός και προφορικός και η γραμμή μας είναι σαφής. Υπάρχει οδηγία για τα, απόβλητα, τα απόβλητα. Δεν είναι παλιά οδηγία είναι μια οδηγία που εγκρίθηκε με συναπόφαση από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο με μια συγκεκριμένη προσέγγιση. Και η προσέγγιση αυτή τι αφορά, αφορά ε, την θέσπιση συγκεκριμένων προδιαγραφών έτσι ώστε τα εξορρυκτικά απόβλητα να διαχειρίζονται με ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την κατασκευή και την διαχείριση εγκαταστάσεων αποβλήτων. Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική πρόληψη ατυχημάτων, συγκεκριμένη, συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης τοξικών ουσιών, λεπτομερείς απαιτήσει περί διαφάνειας ε, στην ενημέρωση του κοινού και επίσης αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά το κλείσιμο κάποιου ορυχείου και οικονομικές εγγυήσεις για κάθε εγκατάσταση προτού εκείνη αρχίσει να λειτουργεί. Αυτή ήταν η απόφαση των συνομοθετών οι επιλογές που υπήρχαν, το να δεχτούμε, το να επιτρέψουμε την εξόριξη χρυσουμεκή ανίδια εφόσον πληρούνται όλες αυτές οι προδιαγραφές ήταν ακριβώς ο λόγος για τον οποίο υπάρχει στην οδηγία υπάρχουν στην οδηγία σαφείς διατάξεις σχετικά με τις συγκεντρώσεις και ανιδίων Εάν ο συνομοθέτης θεωρούσε πως η τεχνολογία αυτή ήταν, δεν ήταν ασφαλής τότε, θα είχαν συμπεριληφθεί σχετικές διατάξεις στην οδηγία για τα εξορρυκτικά απόβλητα όσον αφορά τα όρια συγκέντρωσης ανιδίων. Και εδώ η επιλογή ήταν των συνομοθετών. οι συνομοθέτες δεν χρησιμοποίησαν και κάτι, κάποια εξαιρετικά πρωτότυπη τεχνική. Και αληθεύει επίση ότι για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τα όρια, τα ανώτατα όρια συγκέντρωσης είναι 26 μέρη ένα εκατομμύριο. Για τις εγκαταστάσεις αυτές, το όριο συγκέντρωσης θα είναι 10 μέρη ανά εκατομμύριο το Μάιο του 2018. Για τις νέες εξορρυκτικές εγκαταστάσεις, το όριο συγκέντρωσης είναι ήδη 10 μέρη ανά εκατομμύριο. Τώρα η κυρία Χάση, η κυρία Αντωνέσκου, η κυρία Κλάς ε, ε να ερωτήσεις για το θέμα στη Ρώσια Μοντάνα. Να σας πω κάτι που γνωρίζετε ήδη. Η εξουσία έγκριση σε μια εξοριστική εγκατάσταση βρίσκεται στα κράτη-μέλη, στις εθνικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ελέγχει εάν πληρούνται οι τις οδηγίες και αυτό ακριβώς κάνουμε. Έχουμε ζητήσει να λάβουμε πληροφορίες από τις ρουμανικές αρχές μέσω του πιλότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει εγκριθεί ακόμα το πρόγραμμα αυτό, όμως εμείς ε, προς το παρόν συλλέγουμε πληροφορίες ακριβώς για να ελέγξουμε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και αν υπάρχει συμμόρφωση με την οδηγία για τα εξορρυκτικά απόβλητα. Αυτό το αίτημα έχει σταλεί στην Ρουμανία. Δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση. Φοβάμαι λοιπόν ότι σε αυτό το στάδιο δεν μπορώ ακόμα να σας δώσω κάποια οριστική εκτίμηση του αν το project αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία ή όχι. Τώρα, όπως είπα και στην παρουσίασή μου, υπάρχει μια μελέτη που έχουμε εκπονήσει και με τα χαράς να σας μοιράσουμε αντίγραφα ή κατ' σύνδεσμο. Μπορείτε να βρείτε τη μελέτη και στον ιστοτοπό μας. Πιστεύω πως ανέφερα ήδη ότι αυτή η μελέτη που εκπονήθηκε το 2010 δείχνει ότι καταρχάς εναλλακτικές οι εναλλακτικέ ε, λύσεις στην εξόριξη χρυσού μεκιανίδια δεν είναι οικονομικά βιώσιμες. Επίσης η μελέτη αυτή καταδεικνύει ότι καταδεικνύει μάλιστα ότι πολλές φορές είναι περιβαλλοντικά πιο επιζήμια οι εναλλακτικέ τεχνικές εξόριξης. Νομίζω πως απάντησα σε, στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις ερωτήσεις σας, στα κυριότερα ζητήματα που φίξατε τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και θα φροντίσω τα μέλη της Επιτροπής να λάβουν ένα αντίγραφο της μελέτης μας για την εξόρυξη χρυσού μεκιανίδια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με αυτό φτάσαμε στο τέλος της συζήτησης. Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους καλό βράδυ. Αύριο στις 10 θα τα πούμε πάλι και οι συντονιστές παρακαλώ να έρθουν από τις 9. Επίσημα αρχίζουμε στις 10 με τον κύριο Σπρένιερ από την ECTC ε και μετά με τον Επιτροπο όπου θα διεξαχθεί μια ανταλλαγή απόψεων. Καλό βράδυ.